Okay. Good evening. Καλησπέρα. Ας ε, ξεκινήσουμε γιατί δεν έχει μείνει χρόνος. Οπότε, ε, για να γίνει μια σωστή συζήτηση, καλό είναι να ξεκινάμε. Το πρώτο θέμα η έγκριση ημερήσιας διάταξης. Ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Βέρναρ Χόιερ και να δώσω τον ε, λόγο στον κύριο Φανόβερφελτ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τον πρόεδρο Χόιερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ε, συνάντηση αυτή που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τον ρόλο και την συνεισφορά της Τράπεζας στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης Γενικώ, και ειδικώ όσον αφορά το νέο πράσινο deal. Ε, είχε κολλήσει την κίνηση ο κύριο Χόιρ, οπότε 9.30 ώρα τελειώνουν οι διερμηνείς, οπότε θα επιμείνω στο πρόγραμμα, θα είμαι λίγο αυστηρός, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χόιρ για μια εισαγωγή 7 λεπτών και μετά θα εργαστούμε με τετράλεπτα Οπότε όσο πιο μακροσκελής ερώτησή σας, τόσο πιο σύντομη θα είναι αναγκαστικά η απάντηση του κυρίου Χόιρ και θα επιμείνω σε αυτό. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε σε 9.30. Λοιπόν, κύριε Χόιερ, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Καλή χρονιά σε όλους και πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση, δεν το συνηθίζω, αλλά ερχόμαστε από την ορκομοσία της Νέας Κομισιόν ε, στο Λουξεμβούργο, στο δικαστήριο και ε, είχε φοβερή κίνηση, η Επιτροπή ακόμα στο δρόμο είναι. Να ευχαριστήσω τους δύο συμπρόεδρους για την πρόσκληση σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων πως είναι μια τέλεια ευκαιρία με το νέο έτος και δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε με το πί, το νέο πράσινο deal, το InvestEU και τα μεγάλα ζητήματα του κλίματος. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κορμάν, τον εισηγητή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την συνεργασία και αναμένω την περαιτέρω στενή συνεργασία μας στους επόμενους μήνες. Εκτιμώ ιδιαίτερος ε, την στήριξη που παρέχεται στην ε, ΤΕΠ ως ε, Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζεται τον ρόλο μας ως καταλήτη επενδύσεων και για την χάραξη νέων πολιτικών εντός και εκτός της Ένωσης. Και εκτός της Ένωσης το τονίζω αυτό, γιατί η στήριξή σας είναι η μόνη εγγύηση που έχουμε για τις δραστηριότητες μας εκτός της Ένωσης. 60% των οποίων και ακόμη περισσότερο ε, σχετίζονται με το κλίμα. Οπότε για να επιτύχουμε τους ε, κλιματικούς μας ε, στόχους, στους οποίους λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε, είναι αναγκαίο ακριβώς να τονίσουμε την εγγύηση που μας παρέχεται μέσω του προϋπολογισμού. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η ΕΤΕΠ και το θηγατρικό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είναι κάτι το οποίο συμφέρει τους ε, φορολογούμενους, καθώς κινητοποιεί και ιδιωτικά κεφάλαια. Να σα αναφέρω ένα ενδεικτικό αριθμό. Έχουμε ένα καταβεβλημένο κεφάλαιο 17 δισεκατομμυρίων ευρώ. ευρώ. Συν τα αποθεματικά που έχουμε συσσωρεύσει. Το καταβεβλημένο λοιπόν είναι 17 δισεκατομμύρια μόνο. Έχουμε έναν ισολογισμό 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μοναδικό όσον αφορά τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και ένα μοναδικό πλεονέκτημα που παρέχουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν πολύ αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς ε, πόρους. Η προστήριξη των πολιτικών που εσείς καθορίζετε και εμείς ακολουθούμε. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal είναι το μεγαλύτερο και τολμηρότερο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Αφορά όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και την συνοχή και καλωσορίζουμε την σύνδεση με ένα μηχανισμό δικαίης μετάβασης που σκοπεύει να σα παρουσιάσει η Κομισιόν αύριο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βασίζεστε στην Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει αποτελέσματα στο Green Deal. Χαίρομαι ιδιαίτερο ε, για το ότι πλέον όλε μου οι προσπάθειε θα εστιάζονται σε αυτό και αναμένουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα ε, από αυτά τα οποία θα σας πει και εσά αύριο η Κομισιόν. Όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά να προσφέρουμε στο μέτωπο του κλίματος. Ίσως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει όλη την τελευταία δεκαετία, αλλά είμαστε ο μεγαλύτερο χρηματοδότης ε, κλιματικών δράσεων εδώ και δεκαετίες σύμφωνα βεβαίως και με τον ηγετικό ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Είμαστε η κινητήρια δύναμη πίσω από τις, ε, την στήριξη των πολυμερών ε, αναπτυξιακών τραπεζών ε, στην Συμφωνία των Παρισίων, αλλά και ο μεγαλύτερος πολυμερής επενδυτής ανά τον κόσμο. Πέρσι είχαμε μια ιστορική στιγμή, ανακοίνωσα την πρόθεση της τράπεζας να σταματήσει να χρηματοδοτεί ε, αμυγός ορυκτά καύσιμα και στην δεκαετία που έρχεται θα στηρίξουμε επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για έργα κλίματος και περιβάλλοντος. Η πιο φιλόδοξη πολιτική ε, δημόσιας χρηματοδότησης οπουδήποτε. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Όταν λέμε ότι θα κινητοποιήσουμε χρηματοδότηση ενό τρισεκατομμυρίου σε βάθο δεκαετία, σημαίνει ότι θα κινητοποιήσουμε, θα μοχλεύσουμε τα χρήματα που θα μα δώσετε εσεί, οι άλλοι, οι κεφαλαίοι αγορέ. Δεν έχουμε ένα τρισεκατομμύριο στα υπόγεια τη τραπεζα έτσι. Γιατί ε, συχνά υπάρχει αυτή η παρεξήγηση και κυκλοφορούν διάφορα διάφοροι αριθμοί απίστευτοι η στόχοι μας είναι σαφείς. Ε, πέρα από την επίτευξη αυτού του τρισεκατομμυρίου σκοπεύουμε να μέχρι το 2025 τα κλιματικά να αποτελούν 50% των δραστηριοτήτων μας. Ε, γιατί βεβαίως δεν έχει νόημα το 50% να πηγαίνει σε κλιματικές δράσεις και με τα υπόλοιπα να καταστρέφουμε το καλό το οποίο κάνουμε με τις μισές μας δράσεις. Οπότε αυτό εννοούμε με την ευθυγράμμιση. Η απομάκρυνση από τον άνθρακα θα, θα απαιτήσει πολύ περιπλοκές προσαρμογές από τους πολίτες και τα επενδυτικά ταμεία και συχνά βεβαίως αυτή είναι αυτή με τους λιγότερους πόρους και οι πιο ευάλωτες περιοχές. Θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μία νέα όθηση στην πολιτική της σύγκλησης. Γι' αυτό ακριβώς ε, θέλουμε την δική σας την στήριξη για να δημιουργήσουμε οικονομική αναζωογόνηση. Δεσμευόμαστε για μια δίκαιη μετάβαση των πιο ευπαθών ομάδων για να μην μείνει κανένας πίσω. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να συνεργαστούμε για ένα μηχανισμό δίκαιη μετάβαση. Να τονίσω όμω επίση πω μιλάμε εδώ για την φιλοδοξία τη Ευρώπη να παίξει ηγετικό τεχνολογικά ρόλο στα του κλίματος πρέπει να είμαστε οι πιο προχωρημένοι στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα μας επιτρέψουν να εργαστούμε με σαφώς χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Κύριε και κύριοι, ε, για πολλού θεωρείται ότι η συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε με το σχέδιο Juncker. Δεν ισχύει όμω αυτό. Συνεργαζόμαστε εδώ και δεκαετίε και πάντα βεβαίω το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μελών του. Όπω είχε πει και ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, τον Ιούλιο του 2018, η Κομισιόν δεν είναι τράπεζα και η τράπεζα δεν είναι η Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα έχει στηρίξει και ακριβώ ζητάει να εστιάσουμε ε, ο καθένα σε αυτό το οποίο κάνει καλύτερα. Αυτό το οποίο κάνει καλύτερα η τράπεζα λοιπόν είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει του στόχου τη μέσω βιώσιμων επενδύσεων. Όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο Juncker το 2015 υπήρχαν πολλέ επιφυλάξει. Η κινητοποίηση 350 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες επιπρόσθετες επενδύσεις, οι περισσότερες από τον ε, ιδιωτικό τομέα, με 21 δισεκατομμύρια εγγυημένο προπολογισμό, 16 από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και 5 από την τράπεζα, δεν πρόκειται να είναι κάτι το εύκολο. Δείξαμε ότι μπορεί να γίνει. Και έτσι μετασχηματίσαμε τον ε, τρόπο χρήσης των δημοσίων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των δημοσίων πολιτικών. Έχουμε κινητοποιήσει περί τα 460 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον και θα έχουμε αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,8% και θα έχει δημιουργήσει το πακέτο αυτό 1,7 εκατομμύρια δουλειές οι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανακάμψει, αλλά η ανάκαμψη είναι άνηση μεταξύ χωρών και κλάδων. Σκεφτούμε παραδείγματο χάρη του ε, τομεί των υποδομών ή της καινοτομία, όπου είναι πίσω η τη καινοτομια οπου Ένωση. Θεωρώ ότι για να είναι επιτυχημένα το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να οικοδομήσουμε στι επιτυχίε μα να συνεχίσουμε με τη φιλοδοξία του σχεδίου Juncker και ελπίζουμε να επιτύχουμε συμφωνία επί του νέου ΠΔΠ σύντομα για να συνδεθεί το σχέδιο η φόρο αναπτύξή ε, με το πρόγραμμα Invest EU. Τα δημοσιονομικά αυτά μέσα λειτουργούν μόνο εάν λάβουμε υπόψη και τι απαιτήσει τη αγοράς. Πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα, να προσαρμοζόμαστε στι απαιτήσει τη αγοράς. Εμείς ακριβώς θεωρούμε ότι θα παίξουμε ένα ρόλο καταλήτη, θα κλείσουμε κάποια κενά εκεί όπου υπάρχουν από την αγορά, εκεί όπου η αγορά είναι αναποτελεσματική. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι για να ανταποκριθούμε στις αλλαγές ε, που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και βεβαίως έχουμε και μία λιτή δομή ε, διοίκησης. Δύο λόγια της δραστηριότητας μας εκτός της Ένωσης. Πέρα από το κλιματικό ζήτημα προβλέπω ότι η ανάπτυξη την οποία ε, την σκεφτόμαστε δυστυχώ μόνο στο πλαίσιο της μετανάστευσης, θα αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γεγονός είναι ότι μέσω της ε, δικής σας τράπεζα η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις ε, παγκόσμιες ε, φιλοδοξίες της. Αναφέρθηκα στην ιστορική ανακοίνωση για τα θέματα της ενέργειας και του δανεισμού και του κλίματος η Ευρωπαϊκή λοιπόν έχει την αναπτυξιακή της τράπεζα, την ΕΤΕΠ, αλλά υπάρχει η εντύπωση που φαίνεται και στην ε, έκθεση της Επιτροπής Σοφών ε, του Τόμας Βίζερ ότι η ε, ΕΤΕΠ αποφεύγει τα ρίσκα. Εμείς όμως κάνουμε αυτά τα οποία μας ζητάτε. Αυτά εφαρμόζουμε και αναλαμβάνουμε τους κινδύνους που μας ζητάτε. Για πάνω από 50 χρόνια η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την εξωτερική αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης σε πάρα πολλές χώρες με ελάχιστο κόστος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις υπήρους. Έχουμε έκθεση σε 43 από τα 59 πιο εύθραυστα ευάλωτα ασταθή κράτη και ε, περιοχές. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία συχνά μιλάνε η πολιτική. Και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την πλήρη συνοχή όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε απέναντί μας στο τραπέζι των οποιονδήποτε Κινέζους, Αμερικανούς, Ιρακινούς. Λοιπόν, εάν θέλουμε να παίξουμε παγκοσμίως ηγετικό ρόλο στην κλιματική πολιτική. Χρειάζεται μια ισχυρή χρηματοδότηση, άρα μια ισχυρή τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζητάω λοιπόν την στήριξή σας στις ε, διαπραγματεύσει για το μέσο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κεντρικό ρόλο της ε, τράπεζάς μας. για να παίξει τον ρόλο που έχει ε, στις δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω εδώ κύριε Πρόεδρε, γιατί μου είπατε να περιοριστώ σε 7 λεπτά. Τα υπόλοιπα θα τα πω στις απαντήσεις. Ε, είπα 7 λεπτά πάνω κάτω. Εντάξει, μιλήσατε λίγο παραπάνω. Θα, θα δούμε. Κύριε Φερνάνδες, Είσαι στο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χόγερ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Το σχέδιο Juncker, το σχέδιο για ε, στρατηγικές επενδύσεις, στέφθηκε με επιτυχία και συμμετείχα ως ε, συντονιστής. Πρόκειται για μια επιτυχία η οποία κινητοποίησε... Διακοπή. Δεν ακούτε τη διερμηνία. Συνεχίζω λοιπόν. Έλεγα ότι ήμουν ευτυχής που ήμουν συνεισηγητή για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το πρόγραμμα InvestEU και τι ρόλο περιμένετε να παίξετε εσείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η Επιτροπή και το Συμβούλιο μίλησαν για 650 εκατομμύρια. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιος θα είναι ο ρόλος τώρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το Ταμείο για να υπάρξει αυτή η δίκαια μετάβαση. Κάτι άλλο τώρα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ακριβώς για τη δίκαια μετάβαση. Πώς θα χρηματοδοτηθεί. Προβλέπουμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ το InvestEU με 75% εγγύησης από την ΕΤΕΠ και μετά ποιο θα είναι το ποσό που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κινητοποιήσει ώστε να συμμετάσχει και αυτή στο μηχανισμό αυτό για τη δίκαια μετάβαση. Και έχω και άλλη μία ερώτηση η οποία έχει να κάνει με την Πράσινη Συμφωνία. Ε, τι ποσοστό έχει προβλέψει η ΕΤΕΠ για την χρηματοδότηση, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ποιος είναι ο ρόλος που επιφυλάσσει στον εαυτό της η ΕΤΕΠ ώστε να συμμετάσχει σε αυτήν τη νέα πράσινη συμφωνία που πρότεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως επίσης, όπως σας ρώτησα πριν, και για τον μηχανισμό δικαίας μετάβασης το ίδιο. Ναι, ε, αν νόμιζα ότι θα ακούγα περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, θα απαντήσω, ναι. Τι μάθαμε από την εμπειρία μας με το σχέδιο Juncker. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα για το Invest EU. Δηλαδή, ό,τι λειτουργήσε καλά, να το κρατήσουμε, ό,τι δεν πήγε αρκετά καλά, να διορθωθεί, να προσαρμοστεί. Όταν ξεκινήσαμε με την ιδέα αυτή για το InvestEU, αυτό έγινε σε δύο βάσεις, απλοποίηση και streamlined. Εγώ θα φροντίσω ε, να υλοποιηθούν αυτές οι δύο ιδέες. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολη η απλοποίηση, μερικές φορές οδηγεί σε μεγαλύτερες περιπλοκές, αλλά θα το φροντίσουμε. Έπειτα, το InvestEU θα πρέπει να επικεντρωθεί στις κύριε επενδυτικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να ξεπεράσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις ή τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών στόχων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, έχουμε ένα στόχο κλειδί που είναι η σύγκληση, η συνοχή από τη μία και η καινοτομία από την άλλη. Μπορεί να αποδειχτεί ξεκάθαρα ότι το πετύχαμε με το σχέδιο Juncker και με τις δραστηριότητες στα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα, εκτός δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χώρες που είχαν ανάγκη από στήριξη για προσχώρηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή για άλλα, χρησιμοποίησαν και την καινοτομία. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας την ιδέα ότι είναι χωριστά αυτά και αντιφατικά μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατεύθυνση που παίρνουμε. Ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα, ε, συνοχή, σύγκληση και να είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την τεχνολογία και να μην σέρνουμε τα πόδια μας. Ωραία. Η κυρία Φερέιρα τώρα είναι η επόμενη. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Χόγερ. Η ΕΤΕΠ όταν ξεκίνησα εγώ την καριέρα μου, ε, η ΕΤΕΠ ήταν το σημείο στο οποίο είχα ξεκινήσει ε, την ε, καριέρα μου εγώ ως μαθη, μαθητευόμενη. Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο μετάβαση σε μια πράσινη τράπεζα που θα εξυπηρετήσει την επίτευξη των στόχων του Παρισιού και ε, μια πιο οικολογική οικονομία. Το περιβάλλον και η κατάστασή του είναι μια απέτηση των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι μία από τις βασικές ανησυχίες των πολιτών σύμφωνα με το τελευταίο ευρωμαρόμετρο. Και νομίζω ότι οι διαμαρτυρίες που ακούγονται μας πρόχνουν στο να πάρουμε πιο ριζοσπαστικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ χρήσιμη η δέσμευση να κινητοποιηθεί ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση και το 50% της χρηματοδότησης ε, θα αφορά το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πολύ συχνά ε, επενδύσεις για το κλίμα και για την ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαιη μετάβαση, κολλάνε. <clears throat> υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα στην αγορά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξή. Ε, τι γίνεται με τα πράσινα ομόλογα, πού βρίσκεται η συζήτηση και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αύξηση των επενδύσεων. Δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος ε, των, ε, τραπε, των απτυξιακών τραπεζών προκειμένου να καλύψουν κενά της αγοράς. Τρίτον, πώς βλέπετε τη σχέση αυτών των τραπεζών με την ΕΤΕΠ σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Καλώς λοιπόν ξανά πίσω θα έλεγα αλλά θα βρούμε μια καινούρια πλατφόρμα συνεργασίας. Και σίγουρα το, το, κλιματικό είναι μια τέτοια πλατφόρμα. Ε, τις τελευταίες ε, τρεις δεκαετίες έχουμε δει σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, πτώση του τείχους του Βερολίνου ο πόλεμος του Ιράκ η 11η Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι το πολύ βασικό θέμα της συνειδητοποίηση του περιβαλλοντικού προβλήματος ε, πέρσι είναι στο ίδιο επίπεδο σημασίας με αυτά τα τρία. Ε, συναντήθηκα σε μια εκδήλωση τον Απρίλιο με τον πρόεδρο της ε, Γερμανίας για να ευχαριστήσουμε οργανώσεις νέων, μη πολιτικές οργανώσεις, μη κομματικές οργανώσεις ε, νέων για την ε, συνδρομή τους την συνειδητοποίηση του κόσμου κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών. Είναι λοιπόν να, δυνατόν να κινητοποιήσουμε τους νέους ε, και αυτό είπα στον πρόεδρο και συμφώνησε και αυτοί οι νέοι θα μας κινητοποιήσουν και εμάς και αυτό είναι κάτι μόνιμο. Τώρα, έχουμε διάφορα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να γίνει και φιλική προς επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και με τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες γιατί μόνο μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε με αυτές. Ο κόσμος ε, μας χρειάζεται γιατί οι αγορές έχουν αποτύχει προς το παρόν και θα πρέπει να επενδύουμε όλοι μαζί. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Εννοείται ότι όσο πιο σύντομε είναι οι ερωτήσει σα και οι παρατηρήσει σα, τόσο περισσότερο χρόνο έχει ο κύριο Χόγερ για να απαντήσει, έτσι. Τέσσερα λεπτά είναι τέσσερα λεπτά. Ο κύριος Χένα Λουόμα, παρακαλώ τώρα. Πρόεδρε Χόγερ, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ και πάλι. Και εγώ έχω κάποια εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πριν από 10 χρόνια ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να σας πω ότι η τράπεζα έχει αλλάξει παντελώς τώρα. Κάτι που είναι θετικό. Η τράπεζα όντως παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της. Η Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο Juncker αποτελούν τέτοια παραδείγματα επιτυχίας. Συγχρόνως όμως, καθώς επεκτείνεται ο ρόλος της τράπεζας αυτής, ε, πρέπει να κοιτάμε όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα και να είμαστε σίγουροι ότι ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επιπλέον χρήματα που πηγαίνουν εκεί όπου η αγορά δεν τα καταφέρνει, εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και όχι να αντικαθιστά ιδιωτικές επενδύσεις. Οπότε ρωτάω, μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι η χρηματοδότηση προγραμμάτων, σχεδίων από την ΕΤΕΠ όντως είναι επιπλέον χρήματα και τι κριτήρια χρησιμοποιείτε για να καταλήγετε σε αυτό το συμπέρασμα. Επίσης, βλέπετε να χρειάζεται καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τους στόχους, τους περιβαλλοντικούς και τους αναπτυξιακούς. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. δεύτερη, για τις αλλαγές που γίνονται. Η δικιά μου ομάδα στηρίζει απόλυτα την ιδέα να γίνει κλιματική τράπεζα η ΕΤΕΠ. Μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι και η κοινωνική διάσταση θα συμπεριληφθεί. Και στο μέλλον θα χρηματοδοτεί την υγεία, την εκπαίδευση, ώστε να υπάρχουν ίσες συνθήκες για όλους. Όταν γίνονται αλλαγέ, τέτοιοι στόχοι μερικές φορές ξεχνιούνται. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλό που συζητάμε αυτό το θέμα, την κοινωνική διάσταση, αλλά και το θέμα του crowding in and crowding off. Η πεποίθησή μου είναι ότι ένα δημόσιο όργανο όπως είναι η, Ευρωμα... η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν πρέπει να αντικαθιστά ιδιωτικές επενδύσεις. Αν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να κάνει επενδύσεις, να τις κάνει. Και οι δημόσιες επενδύσεις το ίδιο. Αλλά υπάρχουν κενά, υπάρχουν λήψεις, όπου μπορεί να καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα. Με σαφή κριτήρια μπορούμε να δείξουμε ότι η αγορά δεν θα τα έχει καταφέρει. Βέβαια, μερικές φορές ακούμε επικρίσεις ότι δεν αφήνουμε τις ιδιωτικές τράπεζες να επενδύσουν και παρεμβαίνουμε εμείς. πρέπει να δούμε γιατί έρχεται κανείς σε μας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τράπεζάς μας είναι ότι είμαστε μια τράπεζα με επιστήμονες, μηχανικούς, ίσως και περισσότερο από ό,τι τραπεζίτες θα έλεγα. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς γνωμοδοτούμε ή συμβουλεύουμε, γνωμοδοτούμε για τεχνολογικά περίπλοκα ζητήματα, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι στη γνωμοδότησή μας. Και έτσι πολύ συχνά καταλήγουμε ε, σε συμπεράσματα για κάποιο περίπλοκο ε, σχέδιο και τον κρίνουμε και μετά έρχονται η... έρχεται ο ιδιωτικό τομέα και λέει μπορούμε και εμείς να συγχρηματοδοτήσουμε γιατί αφού λέτε ότι είναι καλό γιατί να μην συμμετέχουμε κι εμείς. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί επ' αυτού γιατί όπως είπα και στην αρχή τα χρήματα που έχουμε, τα 70 εκατομμύρια είναι από εμά και τα υπόλοιπα έρχονται από τι αγορέ που δεν σα δίνουν 70-90 εκατομμύρια κάθε χρόνο ομόλογα αν δεν ε, χρησιμοποιήσετε εσεί τα χρήματα με σοφό τρόπο. Έπειτα, ε, είμαστε επιτυχεί τα τελευταία χρόνια με τα πράσινα ομόλογα, οπότε σκοπεύουμε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση με τα ομόλογα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα συνεχίσουμε με το νερό, με την υγεία, ε, με την εκπαίδευση, γιατί πρέπει όντως να υπάρξει περισσότερη κινητοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ευχαριστούμε κύριο Σούστερ, έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω χαιρετίζω το ότι θα μετασχηματιστείτε σε μια κλιματική τράπεζα, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις για το πώς θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, ε, είπατε ότι 50% θα πρέπει να πάει σε επενδύσεις που θα προστατεύουν το κλίμα. Με ποια κριτήρια θα ε, δίνονται οι άλλες, θα γίνονται οι άλλες επενδύσεις για να μην είναι ευλαπτικές. Ε, απλά θα αποκλείονται τα ορυκτά καύσιμα ή υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Θα συνεχίσετε να προωθείτε αεροδρόμια παραδείγματο χάρη και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία δεν είναι ουδέτερα προς το κλίμα. Δεύτερον, πολλές επενδύσεις απαιτούνται στον ε, δημόσιο τομέα, στο επίπεδο των ε, δήμων ή περιφερειών. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και συχνά μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης. Πώς θεωρείτε ότι θα το καταφέρετε αυτό και ειδικά με τις ε, επιχειρήσεις οι επενδύσεις ε, των επιχειρήσεων δεν είναι πάρα πολύ αποδοτικές με την ε, παραδοσιακή ε, έννοια. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε παραπέρα και από το σχέδιο Juncker στο τι θα χρηματοδοτήσετε. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά την ε, ικανότητα αναχρηματοδότησης της ε, ΕΤΕΠ, γιατί βεβαίως αυτό εξαρτάται και από το πώς αξιολογείται και η δική σας ε, πιστοληπτική ικανότητα και εκεί πέρα η διατήρηση του 3α είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση. Βεβαίω το 3α τη τράπεζα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμά. Αν δεν το προστατεύσουμε, θα γίνει τα πράγματα πάρα πολύ ακριβά για του μετόχου. Και αυτό βέβαια αφορά και εσά. Αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κράτος μπορεί να ζήσει με αξιολόγηση χαμηλότερη από 3α. Μπορεί να είναι κάπω πιο ακριβά τα πράγματα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει. Πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν αξιολόγηση 3α. Αλλά εμεί που έχουμε τόσο λίγο κεφάλαιο και βασιζόμαστε στην στήριξη των ε, κρατών μελών ε, μέσω των εγγύσεων, πρέπει να έχουμε το 3α. Οπότε επαγρυπνούμε ως προς αυτό. Η ευθυγράμμιση τώρα με το Παρίσι είναι συνολική, όπως είπα πριν. Δηλαδή, αν είμαστε ευθυγραμμισμένοι και με τον στόχο του 50%, δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο 50% θα είναι βρώμικα εντό αγωγικών έργα που θα καταστρέφουν ό,τι κάνει το άλλο μισό. Οπότε πρέπει να γίνεται έλεγχος περιβαλλοντικός και κλιματικός για όλα τα έργα, για οτιδήποτε κάνουμε. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στο μεσαίωνα και στο μέλλον θα υπάρχουν αεροδρόμια. Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέμαι πώ χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα αεροδρομίων. Χρειαζόμαστε τόσο πολλά αεροδρόμια. Έχουμε πολλά αεροδρόμια που υπολειτουργούν. Και η τελευταία παρατήρηση. Για τα έργα τα οποία αφορούν καθαρά ορυκτά καύσιμα ή κάτι άλλο. Ε, ως προς αυτό πρέπει να λειτουργούμε ω μια εμπορική τράπεζα, γιατί εάν ω τράπεζα επενδύσουμε σε ένα έργο το οποίο θα έχουμε στον ισολογισμό μα για 35-40 χρόνια και γνωρίζουμε εξ αρχή ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων ή κλιματικής ε, θα πρέπει μετά από 10-15 χρόνια να το ξεγράψουμε, τότε ε, προγραμματίζεις ζημιές. Ε, και αν προγραμματίζει ζημιέ, θα είναι στον ισολογισμό μα μια μέρα. Οπότε πρέπει να το αποφύγουμε. Το να φύγουμε δηλαδή από τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι μόνο ένα στόχο που προκύπτει από το περιβάλλον, είναι και λογική οικονομική κίνηση. Και αυτό φαίνεται από το ότι αν δεν το, δεν το κάνει ε, καμία ιδιωτική τράπεζα, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε και εμεί. Εάν κάποιο θέλει να επιδοτήσει τα ορυκτά καύσιμα, μπορεί να το κάνει, αλλά όχι με τα λεφτά του φορολογούμενου που εγγυώνται την ύπαρξη τη τράπεζα. Σα ευχαριστώ, κύριε Χώση. Καλώς ήρθατε κύριε Χόιρε. Πριν από 30 χρόνια ήμουν μέλο μιας μη κυβερνητική ε, οργάνωσης ε, που κάναμε εκστρατεία εναντίον της ΕΤΕΠ. Ε, τώρα παραδεχόμαστε τη δράση σας για όλα αυτά τα θέματα. Ε, τρεις βασικές λέξεις υπάρχουν εδώ. Η ταξονομία, η ικανότητα και η συνέπεια. Ε, ήταν πολύ σημαντικό να δούμε ότι η πολιτική δανεισμού της ΕΤΕΠ ε, για την ενέργεια επηρέασε ε, την ταξονομία. Σε ποιο βαθμό η ΕΤΕΠ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη νέα ταξονομία ε, στην, στον μελλοντικό δανεισμό. Δεύτερον, η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών. Ε, όπως λέτε και εσείς πρέπει να είμαστε συνεπείς, δεν μπορούμε να λέμε τα μισά πάνε στο κλίμα και τα άλλα μισά καταστρέφουν τα πρώτα μισά. Οπότε η ερώτηση είναι ε, σε ποιους άλλους τομείς θα αναπτυχθούν ε, πολιτικές, θα διαμορφωθούν πολιτικές ε, που θα συνάδουν με την πολιτική για το κλίμα. Για παράδειγμα στις μεταφορές. Οι εκπομπέ ε, αερίων του θερμοκηπίου, για παράδειγμα, θα πρέπει να μα απασχολήσουν πάρα πολύ. Και θα πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τέλο, η τρίτη λέξη κλειδί είναι η ικανότητα. Ε, το capacity, όπως είπατε και εσείς, ε, έχετε εξαιρετικούς εμπειρογνώμονε που βοηθούν στην διαμόρφωση των προγραμμάτων και των σχεδίων. Και εγώ, προερχόμενος από την κεντρική Ευρώπη, μπορώ να σας πω ότι αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ω Κοινοβούλιο για να σα βοηθήσουμε και τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως ΕΤΕΠ για να βοηθήσετε κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίηση με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτετε εσείς. Γιατί εμείς δεν διαθέτουμε επαρκή εμπειρογνωμοσύνη, θα μπορούσατε να μα βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Να απαντήσω για καταρχήν να ξεκινήσουμε με ταξονομία. Ε, όταν ε, ε, δημιουργήσαμε το 2007 τα πράσινα ομόλογα μας χαρακτήρισαν τρελούς, τώρα ε, βλέπουμε την τεράστια επιτυχία που έχουν. Βέβαια, μάθαμε και τα μαθήματά μας, διδαχθήκαμε, γιατί ε, είδαμε πώς μπορεί να είναι επιτυχές και το greenwashing, δηλαδή ε, η, η επιφανειακή οικολογική προσέγγιση και αυτό μας έχει βλάψει. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ό,τι ονομάζεται πράσινο είναι πραγματικά πράσινο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καλωσορίζω την εργασία της ε, Καμισιόν για την ταξινομία. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα η ε, προσπάθεια αυτή είναι πολύ αξιόλογη, γιατί ε, θα μπορούσε να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στον ΩΣΑ. Δεύτερον, θα πρέπει να εξελίξουμε τις πολιτικές μας. Οι μεταφορές, για παράδειγμα, είναι ένας κλάδος κλειδί Γνωρίζετε ότι πάντοτε προηγείται διαβούλευση. Αυτό δεν γίνεται λοιπόν, αυτέ οι αλλαγέ δεν γίνονται εν μία νυχτή, αλλά είναι σημαντικό πράγμα να δείξουμε μια συνέπεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ικανότητέ μα. Η ικανότητα τη τράπεζα είναι πράγματι περιορισμένη. <clears throat> Είμαστε η μεγαλύτερη προφανώ ε, πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα στον κόσμο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε από μόνοι μας να πετύχουμε όλου αυτού του στόχου. Χρειαζόμαστε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, σόφρονες, και να μην υποτιμούμε την ανάγκη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Ε, χρειάζεται λοιπόν να ε, επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα. Και σίγουρα οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης μπορεί να βοηθηθούν από την εμπειρογνωμοσύνη μα, από την τεχνική προνοσή που διαθέτουμε. Οπότε δεν χρειάζονται μόνο χρήματα. Ενδεχομένω τα χρήματα είναι πάντοτε τόσο απαραίτητα, όσο μερικέ φορέ η τεχνική συνδρομή. <clears throat> Και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορεί να βοηθήσει και η Κομισιόν με τη δική μα στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπισλάρου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων εδώ μια τόσο σημαντική στιγμή Αύριο το Σώμα των Επιτρόπων θα εγκρίνει την πρωτοβουλία και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εντάξει, έχουμε ένα σχέδιο και τον μηχανισμό. Με 7,5 δισεκατομμύρια επιπλέον από τον προϋπολογισμό και μετά έχουμε και 45 εκατομμύρια από το InvestEU και μετά έχουμε και τα δάνεια που θα συμπληρώσουν το ποσό. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, ξεκινάτε, με την ε, σύγκληση και την απλοποίηση. Όμως, είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε πώς θα περάσει το μήνυμα ότι υπάρχουν ευκαιρίες ε, κατευθείαν στους παράγοντες της αγοράς. Οπότε η ερώτηση είναι, τις προσπάθειές σας που πρέπει να είναι ουσιαστικές, πώς τις βλέπετε μέσω των αξιωματούχων στις διάφορες χώρες μέλη. Βλέπετε συνεργασία, εταιρική σχέση. Έπειτα, μιλάμε για τα πολυπληθή εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα. Πολλές φορές πάμε και συζητάμε με τον ιδιωτικό τομέα και όταν το έκανα εγώ αυτό, είχα την αίσθηση και τους άκουσα να μου λένε δηλαδή, ότι είναι πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα που συζητάμε και επιμένω στο θέμα της επικοινωνίας γιατί εγώ έρχομαι από μια χώρα και μια περιοχή όπου το ενδιαφέρον των παραγόντων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, είναι πολύ μεγάλο, αλλά διαμαρτύρονται γιατί λένε ότι δεν έχουν αρκετές πληροφορίες. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να είναι διαθέσιμα τα μέσα που εσείς φροντίζετε να είναι, ναι, αλλά έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Πώς το κοινωνάτε αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το InvestEU και είμαι σκιώδη συζητητής για αυτό το θέμα. Συναντήθηκα με πάρα πολλού επιτόπου, μικρομεσέ επιχειρήσεις κλπ. Και χάρηκα πολύ που είδα ότι ένα από τα θέματα που βάζουν για την έλλειψη δεξιοτεχνιών στην αγορά για αυτούς είναι σημαντικό. Και όλοι πιστεύουμε ότι σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η ΕΤΕΠ για την καινοτομία, για την ψηφιακή τεχνολογία, να καλυφθούν τα κενά κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι εσείς θα επικεντρωθείτε στην οικονομική στήριξη όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη. Οι ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές υποδομές θα αποτελέσουν προτεραιότητα για σας και έπειτα θα συμφωνούσατε να επενδύσετε και στα κοινωνικά πέρα από τα 4 δισεκατομμύρια. Άπαξ και φανεί ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Τέσσερα λεπτά περίπου χρησιμοποίησατε. Ε, ναι, αλλά ήταν ε, σημαντικά. Ναι, αλλά η απάντηση του κύριου Χόγκερ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σύντομη. Ναι, λοιπόν, ναι, φυσικά και τα βλέπω όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά οι μελέτες που κάναμε εμείς και σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνούν και με άλλους θεσμούς, το θέμα είναι πού είναι τα εμπόδια. Οι δεξιότητες είναι ένα εμπόδιο. Ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση ικανοτήτων είναι το άλλο. Έχουμε μερικές επιτυχίες σε χώρες μέλη που θέλουν να κάνουν, αλλά δεν τα κάνουν γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τελικά τα διαθέσιμα χρήματα. Και τρίτον, πιστεύω ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά ε, στην ε, ψηφιακή εποχή. Ακόμα και σε εμά νομίζουμε ότι τα ψηφιακά είναι πληροφορική. Αμ, όχι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι κι αλλιώ, εμείς έχουμε τα περισσότερα δεδομένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που υπάρχουν. Δεν τα χρησιμοποιούμε αρκετά. Επιπλέον θα έλεγα ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Πάντα μπορεί κανείς να κάνει περισσότερα. Αλλά όταν εγώ έφτασα στην τράπεζα δεν είχαμε ακούσει πολλά και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και η τράπεζα προβάλλεται περισσότερο Σίγουρα χρειάζεται και οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν και παραγωγή ε, περισσότερη πρόσβαση, μεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Κύριο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα είμαι σύντομο ώστε να μπορέσουν όλοι να ακούσουν τη μετάφραση. Λοιπόν, ε, χαίρομαι που η ΕΤΕΠ μπαίνει στο δρόμο της οικολογικής μετάβασης στον πλανήτη και στον κόσμο. Σας καλώ όμω, παρακαλώ να μην μείνετε στα μέσα του δρόμου, γιατί κατά τη γνώμη μου ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς μέχρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μετατρέψει την ΕΤΕΠ και την έχουμε καταστήσει κλιματική τράπεζα. Αυτή η κλιματική τράπεζα που θέλουμε να έχουμε θα πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και κυρίως όταν οι πιστώσεις της τυχαίνουν διαχείρισης μέσω ενδιάμεσων, τότε η κλιματική τράπεζα πρέπει να εγγυθεί ότι τα χρήματα τα οποία εξοδεύονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσο και εκτός δεν χρηματοδοτούν έργα τα οποία παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη φύση. Αντίθετα, ότι προστατεύουν το κλίμα και γι' αυτό χρειάζεται ένα αξιόπιστο και ξεκάθαρο σχέδιο δράσης. Πότε λοιπόν εσείς θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε ένα τέτοιο σχέδιο δράσης και πότε θα ενημερώσετε τις σα σας πολιτικές κυρίως εκείνης δανεισμού στις μεταφορές και επίσης όσον αφορά τη διαφάνεια. Και επειδή πριν μίλησα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πότε σχεδιάζετε να υιοθετήσετε συνολική και συνεκτική ε, στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα με κυρώσεις όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς θα κινητοποιήσετε μέσα για να προσλάβετε ειδικού για αυτά τα θέματα στην ΕΤΕΠ. Απάντηση. Η φιλοδοξία μας όσον αφορά το κλίμα είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό ίδρυμα ανά το κόσμο. Για μένα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, γιατί ακριβώ τέτοια τράπεζα είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε τέτοια τράπεζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και δίνουμε το παράδειγμα και στις άλλες τράπεζες. Είπαμε 25% κλιματικές δράσεις στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας στην αρχή. Τώρα είμαστε στο 30% και έχουμε σαν στόχο το 50% το 2025. Άρα είμαστε εδώ και καιρό κλιματική τράπεζα και θα το πετύχουμε και αυτό το νέο στόχο. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με το ότι τώρα έχουμε πάρει το όνομα Κλιματική Τράπεζα. Όχι, θα είμαστε Τράπεζα Καινοτομία, Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ε, Τράπεζα Δημιουργία. Και αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Γιατί όταν μιλάμε για δίκαια μετάβαση, μιλάμε για περιφέρειες οι οποίες θα πληγούν όταν εγκαταλείψουν το ρηκτά και πρέπει να βρεθούν νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους αυτούς. Και δεν πρόκειται μόνο για εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, πρόκειται και για την απασχόληση. Γιατί αυτό που δουλεύει στα ορυχεία, ο μεταλλορύχος, δεν ξέρω σε ποια περιοχή τη Ευρώπη. δεν πρόκειται μέσα σε ένα-δύο χρόνια να ξεπεράσει και να βρει καινούργια δουλειά. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε συνολικά. Είναι ένα πακέτο. Εννοείται ότι το κλίμα παίζει ένα ρόλο κλειδί και μας καθοδηγεί στην σκέψη μας, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον κόσμο και άρα να φροντίζουμε για την καινοτομία και την τεχνολογία. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για την έλλειψη αποκλεισμών από οτιδήποτε άλλο. Και να το έχουμε αυτό υπόψη μας κάθε φορά που μιλάμε για πολιτικές αλλαγές, είτε πρόκειται για τις μεταφορές είτε αλλού. Συμφωνώ μαζί σας ότι το θέμα επήγει. Ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Γκίγκολτ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να σας ε, συγχαρώ για τα όσα επιτύχατε στην πολιτική δανεισμού της ε, τράπεζας ενάντια στην αντίσταση της ε, κοινή μας χώρας, της κοινή μας Είναι πολύ θετικό αυτό το ότι έχουμε μεγαλύτερη συνοχή στο κλιματικό μέτωπο και κάτι περισσότερο από συνοχή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω για ένα άρθρο της Financial Times ε, στις 15 Ιουλίου 2019 που προκάλεσε αίσθηση και εκεί πέρα αναφερθήκατε μέσω ε, στο μεγάλο ζήτημα το οποίο άρθρο είχε τίτλο «Ο κρυφός γίγαντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων». Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων είναι τεράστια, έχει μία αξιολόγηση 3α, αλλά έχει ελάχιστε ζημιές. Οι συνολικέ προβλέψεις για ζημιές από δάνεια επί μία δεκαετία ήταν 0,1% σύμφωνα με το άρθρο ε, για το σύνολο των δανείων μακράν το χαμηλότερο ποσοστό των, από τις άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Και κάπως εσείς θέτε γι' αυτό, γιατί όπως είπατε, ε, βεβαίως εσείς αναλαμβάνετε τους κινδύνους που σας ε, ζητάμε εμείς και η ΕΤΕΠ έχει περιορισμένα δικά της ε, κεφάλαια, οπότε αναρωτιέμαι και ρωτώ και εσάς, θεωρείτε ότι η ΕΤΕΠ ε, για να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν όσον αφορά την υλοποίηση του πράσινου deal θα πρέπει να έχει υψηλότερο κεφάλαιο. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δώσουν περισσότερα κεφάλαια όπως κάναμε μετά την μεγάλη οικονομική κρίση για να γίνει πιο εύκολο για την ΕΤΕΠ να αναλάβει τον κίνδυνο που πρέπει για να υπάρξει καινοτομία γιατί η καινοτομία συνοδεύεται από κινδύνους και χρειάζεται και η ΕΤΕΠ ε, να μπορεί να, να λάβει περισσότερους κινδύνου χωρίς να διακινδυνεύει το 3α. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ να απαντήσω. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να το δείτε και από τεχνική σκοπιά, τραπεζική. Έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο λιγμών που έχουμε. Το καταστατικό μας ε, περιορίζει σε ένα λόγω μόχλευση σε 2,5. Δηλαδή δεν πρέπει να δανείζουμε πάνω από 2,5 φορέ το κεφάλαιο που έχουμε. Και το έχουμε σχεδόν εξαντλήσει πλήρω. Και όταν το υπολογίζουμε αυτό, ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζουμε το ρίσκο του κάθε έργου της ε, τράπεζας. Ε, το αν θα αναλάβουμε υψηλότερο κίνδυνο που συχνά απαιτείται όταν μιλάμε για καινοτομία και να δώσουμε εκεί πέρα περισσότερο κεφάλαιο και να μειωθεί το περιθώριο δανεισμού που έχουμε. Κοιτάξτε, όταν ήρθα στην τράπεζα πριν από 8 χρόνια, καταφέραμε, καταφέραμε να έχουμε μια πρώτη σοβαρή αύξηση κεφαλαίου ε, και ακούω αριθμούς ε, για 5 ή 8 ε, δισεκατομμύρια ενέσεις ρευστότητα στην τράπεζα. Βεβαίως τα καλωσορίζουμε, θα μας βοηθήσει λίγο. Θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο <clears throat> εάν πέρα από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια θα είχαμε μία αύξηση στο κεφάλαιο το οποίο πέρα από το κάβαλο το οποίο μας εγγυώνται τα κράτη-μέλη. Οπότε Εντάξει, δεν πηγαίνω συχνά στους μετόχους και λέω χρειαζόμαστε νέο κεφάλαιο, αλλά όπως σας είπα, περισσότερο και από μετρητά χρειαζόμαστε περισσότερες εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη. Αυτά ήθελα να ακούσω, λέει ο κύριος Γκίγκολ. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Ζόγκα. Ευχαριστώ. Η ΕΤΕΠ μέχρι τώρα ασχολείται με χρηματοδότηση καινοτομία, το περιβάλλον, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και την ανάπτυξη των υποδομών. Η ερώτηση μου είναι εξή. Περιμένετε ότι μερικοί από αυτού του κλάδου θα επηρεαστούν από τι αλλαγέ αυτέ που έχετε αποφασίσει. Και δεύτερη ερώτηση για τη χρηματοδότηση υποδομών. Για παράδειγμα, μεταφορές, ή δρόμοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, που έφτασαν, ε, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα ε, και έχουμε πολλά διασυνοριακά σχέδια, στο παρελθόν τουλάχιστον. Τι θα γίνει με αυτά, τι θα γίνει στο μέλλον με τέτοιου είδους σχέδια. Τέλος, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης Προφανώς ε, έχει εξάψει το ενδιαφέρον. Ορισμένες, από τις περιφ... Ορισμένες περιφέρειες θα λάβουν περισσότερη στήριξη προφανώς, έτσι δεν είναι. Η ερώτηση είναι με ποια κριτήρια θα αποφασιστεί η χρηματοδότηση αυτών των περιοχών και για τι είδους ποσά μιλάμε. Ποιες περιφέρειες τέλος πιστεύετε θα είναι επιλέξιμες καταρχήν στο πρώτο κύμα. Απάντηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό θα ήθελα κι εγώ να <laughs> είχα μια πραγματικά αξιόπιστη απάντηση σε όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο ακόμα. Ε, συζητούσαμε την Κομισιόν σήμερα κατά τη διάρκεια τη ορκομοσία τη και μίλησα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαντ, και νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα να εξορροπήσουν αυτό που θα σα παρουσιάσουν τι επόμενε μέρε. Σίγουρα, ε, 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι το Ταμείο της Δίκαιης μετάβασης, ο μηχανισμός αυτός, ε, μαζί με το InvestEU 45 δις. Δεν έχω όμως οριστικά νούμερα. Το σημαντικό είναι πρώτον να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητε τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει το όλο σύστημα αυτό πιο ελκυστικό για τα διασυνοριακά σχέδια. Αυτό αφορά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη σχέση με τις χώρες γειτονίας, για παράδειγμα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, μπορεί να έχουμε εξαιρετική κατάσταση σε ορισμένα από αυτά τα κράτη εσωτερικά, αλλά δεν κάνουν τίποτα συνεργατικά μεταξύ τους. Η Κομισιόν είναι πάρα πολύ φιλόδοξη από ό,τι φαίνεται και αν στηρίξει επαρκώς τις εγγυητικές, εγγυοδοτικές δραστηριότητες της τράπεζας μπορούμε να κάνουμε πολλά. Προφανώς θα είμαστε, η απόδοσή μας θα διαφέρει από χώρα σε χώρα, θα πρέπει να εστιάσουμε όμως στις χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν αρνητικά από τις αλλαγές στην κλιματική ενεργειακή πολιτική. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί αυτή η ισορροπία ακόμα. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο τώρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναφερθώ στο θέμα το οποίο σας απασχόλησε περισσότερο το κλίμα. Έχετε γράψει στην έκθεσή σας ότι η ΕΤΕΠ εγγυάται την κλιματική ουδετερότητα του δανεισμού. Με ενδιαφέρει πώς θα το κάνετε αυτό, πώς το εγγυάστε και πώς καθορίζεται η κλιματική ουδετερότητα και τα κριτήρια τα οποία έχετε αναπτύξει για αυτό. Είναι εμπειρικά, επιστημονικά ή είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί αυθαίρετα, όπως και οι τιμές τις οποίες θέλετε να τηρήσετε. Μιλάμε για ένα... Μια πρωτογραφή που θα ρίχνει τα 550 γραμμάρια ε, διοξιδίου του άνθρακα ανά κιλοβατόρα στα 250 και έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις εν ολίγης για το εάν μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια εκείνη η οποία εκπέμπει λιγότερο, την πυρηνική ενέργεια. Θα στηρίξετε την ε, πυρηνική ενέργεια στον δανεισμό σας, στις επενδύσεις σας. Ε, και αν ναι, πώς ε, σκοπεύετε να επιτύχετε τις ε, φιλόδοξες αυτές μειώσεις διεξιού του άνθρακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο ανοίγεται, γιατί πρέπει να μπούμε σε επιστημονικές λεπτομέρειες. Και δεν θα ήθελα τώρα να φάω ολόκληρη τη συνέδρια. Κοιτάξτε, χρειάζονται σαφή κριτήρια, αλλά Βεβαίω το όριο το οποίο είχε τεθεί για τα 550 γραμμάρια ένα κιλοβατόρα ε, δεν ε, ανταποκρίνεται πλέον σημερινή πραγματικότητα. Μπορούμε να επιτύχουμε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Οπότε, όσο είναι κάτι τόσο απλό, με απλέ τεχνολογίε, να εξακολουθούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, όπω παράδειγμα χάρη με το αέριο. Και μπορούμε να δώσουμε κίνητρα ε, για να φύγουμε από τις παλαιότερες τεχνολογίες. Πρέπει να το δούμε λοιπόν και από μια άλλη σκοπιά. Πώς μπορεί η Ευρώπη να παίξει ηγετικό ρόλο στις ε, τεχνολογίες οι οποίες θα οδηγήσουν αυτές τις εξελίξεις. Ε, γιατί οι άλλοι θα μας ξεπεράσουν. Αν δούμε την Κίνα παραδείγματος χάρη. Όταν οι Κινέζοι λένε ότι θέλουν να κάνουν αυτήν την μεταβολή περί το 2030. Κοιτάξτε, θα το κάνουν. Οπότε πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε και πρέπει να έχουμε υψηλότερες ε, φιλοδοξίες. Και βεβαίως, εντάξει, ομολογώ ότι υπάρχουν ε, τεχνολογικές ε, δυσκολίες και είμαι, σε, διατεθειμένος να σας φέρω σε επαφή με τους ειδικούς μας που μπορούν να τα εξηγήσουν αυτά πιο επιστημονικά. Απλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε πιο φιλοδόξοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζουβέν τώρα. Πρόεδρε, Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας. Έχω δύο ερωτήσεις, παρακαλώ. Πρώτον, για ένα θέμα που ακούστηκε. Για μένα πράσινο σημαίνει γεωργία. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο αγροτικός τομέας, ότι πολλές φορές ε, η βιομηχανία παρεμβαίνει και καταστρέφει τη γη την υγεία των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες επιφάνειες, τις υγρές, τα δάση που βοηθούν γιατί απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα. Από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι η αγροτική γη στοιχίζει σε επενδύσεις κυρίως τα πρώτα χρόνια. Οπότε ρωτάω, είναι μέρος των σχεδίων σας να χρηματοδοτήσετε ή να συνεισφέρετε στην μετατροπή της γεωργίας. Δεύτερον, πιο σύντομα. Η ελευθερία ε, κίνησης ε, υπηρεσιών, τα κτλ. οδηγεί στην απορρίθμιση του κλίματος και ένας φόρος για την εισαγωγή άνθρακα ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει. Και κάτι άλλο θα ήταν η μεταφορά των βιομηχανιών. Όταν βρίσκονται στον ευρωπαϊκό χώρο και τηρούν τους κανόνες, σίγουρα εκπέμπουν λιγότερες ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εσείς θα φροντίσετε για τη μεταφορά των βιομηχανικών ε, δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο χρειάζεται η επικρατεία μας. Απάντηση. Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι όντως χωρίς να χρειάζεται έχουμε επιπλέον εκπομπές. Φυσικά και θέλουμε την πράσινη γεωργία. Βεβαίω και θέλουμε εναλλακτικέ λύσεις. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί Ό,τι είπε ο Γιούνκερ το 2018 ισχύει ότι η Επιτροπή δεν είναι τράπεζα και η τράπεζα δεν είναι η Επιτροπή. Οπότε μην μπερδεύουμε τους ρόλους. Εγώ περιμένω από τους πολιτικούς ηγέτες, από εσά, από τις κυβερνήσεις, από την Επιτροπή να θέσετε τους στόχους και εμείς μετά θα φροντίσουμε να τους χρηματοδοτήσουμε. Μπορείτε να με ρωτήσετε τι πιστεύω εγώ για την πυρηνική ενέργεια. Ωραία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Γιατί εγώ χρειάζομαι τις αποφάσεις του Δικαιωτικού Συμβουλίου που θα στηρίξετε εσείς, το Συμβούλιο, η Επιτροπή. Συνεπώς, Αυτές τις ε, πολιτικές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν οι πολιτικοί. Και για να επανέλθω στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια ε, στα πλαίσια του ενεργειακού δανεισμού της τράπεζας. Αλλιώς θα καταλήξουμε σε χάος. Αν ε, δείτε τα αποτελέσματα της διαδικασίας, δεν υπάρχει τίποτα που να καταστούσε αδύνατο από πλευράς κριτηρίων εκπομπών να χρηματοδοτήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Δεν το έχουμε κάνει βέβαια μέχρι τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον, και ούτε σκοπεύουμε να το κάνουμε στο μέλλον. Οπότε τις πολιτικές αποφάσεις δεν τις παίρνουμε εμείς. Το θέμα τώρα της ενέργειας και του εμπορίου. Εδώ χρειάζεται διάλογος βέβαια. Το θέμα της μεταφοράς των βιομηχανιών, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί αλλά πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια τη αναπτυξιακή πολιτική. Οπότε βέβαια εδώ το εμπόριο πηγαίνει προ την αντίθετη κατεύθυνση ακριβώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριο Παπαδημούλης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Χόγερ, ακούγεται ωραία η εξαγγελία να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων σε μια τράπεζα για το κλίμα. Όπως επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούσαμε ωραία και την εξαγγελία της Κομισιόν για ένα Green New Deal. Αλλά πριν από λίγο μας είπατε ότι περιμένετε κι εσείς να αποσαφινιστούν κάποια μεγέθη από τους πολιτικούς, δηλαδή από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο κτλ. Η ερώτησή μου είναι, επειδή συζητάτε μαζί τους, πότε πιστεύετε ότι θα έχουν αποσαφινιστεί αυτά που σας είναι απαραίτητα για να βάλτε σε εφαρμογή το δικό σας σχέδιο. Δηλαδή, πόσα, γιατί και εκεί δεν συμφωνεί το Συμβούλιο με την Κομισιόν ε, και πώς επίσης θα προστατεύσετε αυτά τα χρήματα που θα τα μοχλεύσετε από το greenwashing, από το να πάνε σε λάθος κατευθύνσεις, σε fake πράσινες πολιτικές. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα. Και μια τρίτη ερώτηση, για να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Η κοινωνική διάσταση, το πώς δεν θα μείνει κανείς πίσω το Just Transition Fund είναι ένα εργαλείο. Με τους σπόρους που διατίθενται είναι επαρκές. Ας βάλουμε μαζί και τα, τους σπόρους από το InvestEU. 45 δις είναι επαρκή για μια δίκαιη μετάβαση ή αυτή η κλιματική στροφή η θετική θα μεγαλώσει τις ανισότητες κοινωνικές και περιφερειακές. Και τέλος, είπατε ότι είναι καλοδεχούμενη μια αύξηση των εγγυήσεων κεφαλαίου από τα κράτη-μέλη. Εσείς σήμερα εδώ θα τη ζητούσατε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να την ζητήσει και να τη στηρίξει. Εσείς μιλάτε τώρα με τους πολιτικούς που είναι άμεσα εκλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως ζητάει από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα κεφάλαια που δίνουν ως εγγυήσεις σε εσά για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Φοντερ Λάιν και οι συνάδελφοί της ανέλαβαν πριν από λίγες εβδομάδες έχουν ανοίξει, θα έλεγα, καινούργια παράθυρα και ε, φυσάει φρέσκος αέρας όρισε κάποιου χοντρικού στόχους η κυρία Φοντερ Λάιν, οι οποίοι πρέπει να διευκρινιστούν βεβαίω. Αυτό χρειάζεται χρόνο και συνεργασία με εσά και με άλλους. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και μπορούμε να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο. Τώρα, εάν οι πολιτικοί ηγέτε της Ένωσης πούν το τι θέλουν να κάνουν και να μας δώσουν για να μπορέσουμε να το πολλαπλασιάσουμε, τότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και όσον αφορά τη μόχλευση, νομίζω ότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Ε, είμαι αισιόδοξο. Για το greenwashing. Ε, είχαμε την εμπειρία μετά το 2007, όταν σε διάφορες ε, τράπεζες έπαιρναν ένα κομμάτι χαρτί, το έδωσαν πράσινο και λέγανε αυτό είναι πράσινο ομόλογο. Όχι, πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια, υπάρχει η ταξονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όρισαν κάποιες αρχές, μια ομάδα συγκεκριμένα για τις ε, αρχές ε, για τα πράσινα ομόλογα, που είχε επηρεαστεί πολύ από τους εμπειρογνώμονες της ε, ΕΤΕΠ και καταλήξαμε σε κάποια κριτήρια στα οποία δεσμεύονται όλοι ανά τον κόσμο. Και δεν θα πρέπει τώρα να περάσουμε σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων γιατί θα πληγεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Και έχουμε κάθε χρόνο αγορές ομολόγων μεταξύ 70 και 90 δισεκατομμυρίων. Αν σταματήσουμε να εμπιστεύουμε θα το κλείσουμε, θα το, κλείσουμε το μαζί. Λοιπόν, με ρωτήσετε επίση για το αν επαρκούν τα 45 δισεκατομμύρια. Ε, αν μου δώσετε και περισσότερα, ε, ευχαριστώ. Ε, και μπορώ να πάω βεβαίως στις ε, κυβερνήσεις και να πω δώστε μας ε, λίγο περισσότερο περιθώριο λίγμων. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες πολυμερείς τράπεζες, τις αναπτυξιακές, δεν θα πω δώστε μας μετρητά, αλλά να αναλάβουμε ακριβώς περισσότερη ευθύνη, να αυξηθούν οι εγγυήσει που μας δίνεται. Έτσι θα μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε μόχλευση πολλαπλάσια αυτών των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται για την ε, δίκαιη μετάβαση και το Investigio. Σας ευχαριστώ. Μας, περιμένουν ελάχιστα ε, λεπτά για το Catch the Eye. Ε, Τρία άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριος Κούσμιου. Mm, ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόγερ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το φυσικό αέριο. Είπατε ότι σταδιακά θα καταργηθούν τα σχέδια που βασίζονται στους ορυκτούς υδρογονάνθρακες, στα θεωρητικά καύσιμα, κυρίως βέβαια στον άνθρακα. Πού μπαίνει όμως το φυσικό αέριο σε όλη αυτή την εικόνα. Η ενέργεια από φυσικό αέριο έχει αναγνωριστεί προσφάτως ως οικολογική πράσινη ενέργεια. Ποια θα είναι η δική σας προσέγγιση. We ε, απομακρυνόμαστε από τους ε, αμυγείς υδρο, από τα αμυγή ορυκτά κάψιμα και τη χρηματοδότησή τους. Από την άλλη μεριά όσα σχέδια ε, υπάρχουν και εξελίσσονται αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται μέχρι να, να ολοκληρωθούν. Τώρα αν συγκρίνεται βέβαια το φυσικό αέριο ή το υδρο, ποιημένο φυσικό αέριο ε, με, τα, με τον άνθρακα, ε, σαφέστατα το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο οικολογικό. Παρ' αυτά, το φυσικό αέριο θα παραμείνει ως μεταβατικό καύσιμο. Οπότε εμείς θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα τέτοιο ενδιάμεσο καύσιμο το οποίο θα καταργηθεί σε ό,τι τη χρηματοδότηση τουλάχιστον σε 10-15 χρόνια ή αν θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία ε, ακυρώνοντα, αποφεύγοντα αποφεύγοντας τέτοιου είδου επενδύσεις. Αναγνωρίζω ότι για κάποια χρόνια θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο, αλλά θα πρέπει ε, να ε, αποφύγουμε τη χρηματοδότησή του. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε την διερμηνία, διότι είναι 9.30 ώρα